συμπρόεδρε από την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων, αξιότιμοι προσκεκλημένοι, καλώς ήρθατε στην συνάντησή μας αυτό το απόγευμα που έχει να κάνει με την επιμόρφωση των δικαστών και των ασκούντων νομικά επαγγέλματα. Οργανώνεται από κοινού μεταξύ των δύο επιτροπών μας. είναι η τελευταία συνάντηση πριν από τις πασχαλινές διακοπές βέβαια Λυπάμαι που μπήκε αυτή τη στιγμή, μια τέτοια μέρα. Αλλά τώρα είχαμε χρόνο, γιατί είχαμε και την τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής μας αυτές τις μέρες, οπότε και αυτό οργανώθηκε και αυτή η συνάντηση τώρα. Για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Σήμερα το απόγευμα λοιπόν, πριν περάσουμε στις παρουσιάσεις των ειδικών, Θέλω να σας πω ότι ο χρόνος που έχουμε στη διάθεσή μας για σήμερα θα επιτρέψει μια γενική επισκόπηση του έργου που γίνεται στον τομέα της επιμόρφωσης ε, για δικαστικά ζητήματα. Ξέρετε ότι κάνουμε πάρα πολύ καλή δουλειά γιατί προσφέρουμε κατάρτιση στους δικαστές, στους ασκούντες ε, γενικά νομικά επαγγέλματα, η νομική ακαδημία επίσης. Και χαιρόμαστε πολύ που έχουμε εδώ και το Συμβούλιο Σεβολογράφων και η ΑΣΟ που είναι η υπηρεσία μας ασύλου και αυτή προσφέρει κατάρτιση για θέματα ασύλου. Χωρίς λοιπόν άλλη καθυστέρηση, είμαι εδώ με την συμπρόεδρο που και εκείνη θα βοηθήσει φυσικά και θα αναλάβει την προεδρία σε λίγο μετά από μένα, ναι. Εντάξει, δεν έχουμε ιεραρχία, έτσι. Σήμερα οι δύο επιτροπές νομικών υποθέσεων και ΛΥΜΠΕ είναι ισότιμες. Πρώτα όλα λοιπόν θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Αλεξάνδρα Ζουρσούντερ που είναι διευθυντή στη Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνη. και θα μας παρουσιάσει την ετήσια έκθεση 2016 όσον αφορά την επιμόρφωση για το 2016. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτές, κυρίες περνάνε από επιμόρφωση για το ευρωπαϊκό δίκαιο και πολύ λίγες χώρες έχουν φτάσει στο 5% που ήταν η ποσόστοση. Είναι σημαντικό βέβαια να πούμε ότι δεν χρειάζεται επιμόρφωση για το ευρωπαϊκό δίκαιο από όλο το προσωπικό των δικαστηρίων, γιατί πολλοί ασχολούνται με υποθέσεις που δεν έχουν να κάνουν με το ευρωπαϊκό δίκαιο, άλλοι ασχολούνται με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Πάντως, σε πολλές χώρες το δικαστικό προσωπικό βοηθάει τους δικαστές, άλλες φορές προσφέρει νομική αρρωγή ή άλλες φορές ασχολείται με τις πληρωμές και συχνά κρατούν αρχεία που άλλοτε έχουν να κάνουν με την Ευρωπαϊκή Ένωση, άλλοτε όχι. Η επιμόρφωση λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο πιστεύουμε ότι είναι σημαντική έτσι κι και πρέπει να ενισχυθεί. Ένα άλλο κενό έχει να κάνει με τις γλώσσες στην αρχική κατάρτιση. 50% των νομικών στην αρχή της σταδιοδρομίας τους δύο ή λιγότερες μέρες έχουν πάρει τέτοια κατάρτιση για το ευρωπαϊκό δίκαιο και πιστεύουν ότι αυτό βέβαια δεν φτάνει δεδομένες της σημασίας που έχει το ευρωπαϊκό δίκαιο σήμερα. Άρα εδώ κάτι πρέπει να γίνει. Θα σας πω τώρα και λίγα λόγια για την Ευρωπαϊκή Οικονομική Αρρωγή. Ξέρετε ότι τα χρήματα δεν είναι τα πάντα, αλλά βοηθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, λοιπόν, προσπαθεί όσο μπορεί περισσότερο να ενισχύσει οικονομικά προγράμματα για να στηρίξει τέτοια επιμόρφωση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει φροντίσει και είμαι γνώμων σε εσά γι' αυτό να υπάρχουν τα μέσα για την υποστήριξη τέτοιων προγραμμάτων. 35% του συνόλου του προπολογισμού 14 με 20 πρέπει να πάει στην ε, επιμόρφωση αυτή. 132 εκατομμύρια σε 7 χρόνια που ακούγεται πολύ, αν, αν συγκρίνεται τα χρήματα που πηγαίνουν για άλλους σκοπούς δεν είναι τόσο πολλά. Το δίκτυο τώρα επιμόρφωσης ε, στην Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη έχει αναγνωρίσει ότι έχει υποφεληθεί πολύ, στηρίζει και αυτό την επιμόρφωση σε όλο το δίκτυο και υπάρχουν περισσότερες επιχορηγήσεις με αποτέλεσμα μεγαλύτερη συμμετοχή στις διάφορες δραστηριότητες επιμόρφωσης και θα τα ακούσετε με περισσότερες λεπτομέρειες σήμερα το απόγευμα. Από το 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει κάνει ετησίως έκκληση για επιχορηγήσεις για να στηρίζονται διακρατικά προγράμματα επιμόρφωσης δικαστικών και υπάρχει στήριξη για πολλά και ενδιαφέροντα προγράμματα. Όπως είπε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2011 εξέδωσε μία ανακοίνωση πριν από έξι χρόνια. Τώρα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι έχουμε να κάνουμε με ένα νέο περιβάλλον και νέες προκλήσεις και πρέπει να εντοπίσουμε λοιπόν θέματα πάνω στο οποίο πρέπει να κάνουμε πιο πολλά, κυρίως όταν έχουμε να κάνουμε την επιμόρφωση των ε, νομικών. Βλέπουμε για παράδειγμα ότι υπάρχουν νέα νομικά επαγγέλματα τα οποία εμφανίζονται και άρα πρέπει και τα άτομα αυτά να επιμορφωθούν. Κατά συνέπεια, τώρα σχεδιάζουμε να ενημερώσουμε την στρατηγική μας για την επιμόρφωση στην δικαιοσύνη και πιστεύω ότι θα έχουμε αποτελέσματα σύντομα. Τώρα, σας είπα για τα κενά όταν πρόκειται για το προσωπικό των δικαστηρίων, για τους νέους επαγγελματίες που μόλις ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους. Εδώ χρειαζόμαστε νέα στρατηγική το ευρωπαϊκό δίκαιο παίζει όλο και μεγαλύτερο ρόλο όσο περνά ο καιρό, οπότε έχει τεράστια σημασία να υπάρχει εκπαίδευση και επιμόρφωση στο ευρωπαϊκό δίκαιο και να μην γίνεται αυτή μόνο μία φορά στα δέκα χρόνια. Πρέπει να σχεδιάσουμε τι θα γίνει και μετά το 2020. Θέλουμε λοιπόν περισσότερη επιμόρφωση για τους δικηγόρους και για τους δικαστούς επιμελητές. Τώρα, Πρέπει να εντοπίσουμε και τις απειλές που έχουμε εξαιτία της ριζοσπαστικοποίησης και της τρομοκρατίας. Οπότε διαπιστώνουμε ότι όλο και περισσότερο στην επιμόρφωση να συμπεριλάβουμε και το προσωπικό των φυλακών τους δεσμοφύλακες δηλαδή, γιατί και αυτοί πρέπει να περάσουν από αυτή την επιμόρφωση. Και υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα προγράμματα, μετά μάλιστα τις τρομοκρατικές επιθέσεις του 2015. Μάθαμε πολλά από αυτά. Βέβαια το ποσοστό είναι πάρα πολύ μικρό, άρα πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να κατανοήσουμε καλύτερα το φαινόμενο και να εξετάσουμε περισσότερο την κατάσταση στις φυλακές σχετικά με τους φυλακισμένους για τέτοιου λόγους. Ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι η ηθική, το κράτος δικαίου και ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Είναι και αυτά ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν. Συνεπώς η επιμόρφωση γίνεται και εδώ αναγκαία. Κάτι άλλο πρακτικό είναι η πρόσβαση σε αποδεικτικά στοιχεία ηλεκτρονικής μορφής. Και σε αυτό χρειάζεται επιμόρφωση. Επίσης, οι χώρες μέλη πρέπει να θεωρηθούν περισσότερο, μια που είναι επιμερισμένη αρμοδιότητα η επιμόρφωση στη δικαιοσύνη, άρα πρέπει να συμμετέχουν όλοι και τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και το Συμβούλιο για τη Δικαστική Εξουσία και άλλα θεσμικά όργανα που υπάρχουν στις διάφορες χώρες μέλη. Η πολιτική μας για την ε, δικαστική επιμόρφωση πρέπει να είναι πιο στοχευμένη για να αντιμετωπίσει επίσης και τις ανάγκες συγκεκριμένων χωρών ή ομάδων χωρών. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι one fits all, ότι ένα μοντέλο ταιριάζει σε όλους. Όχι, υπάρχουν διαφορές και το έχουμε δει αυτό και στα αποτελέσματά μας στην ετήσια αξιολόγησή μας από την επιμόρφωση. Άρα πρέπει να στοχεύουμε καλύτερα με συγκεκριμένες στρατηγικές συγκεκριμένες περιπτώσεις στις χώρες μέλη για να είμαστε πιο αποτελεσματικοί. Επίσης δεν πρέπει να επικεντρωνόμαστε μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει σε ένα βαθμό τουλάχιστον να κοιτάξουμε τι γίνεται και στις γείτονες χώρες, υποψήφιες χώρες, ενδυνάμει υποψήφιες χώρες που ετοιμάζουν μεταρρυθμίσεις στη δικαιοσύνη τους. Δεν λέω ότι είναι ο στόχος της δικιάς μας επιμόρφωσης, αλλά καλό θα ήταν να δούμε τι θα μπορούσαμε να κάνουμε και για αυτούς για να ανταποκριθούμε και στις δικές τους ανάγκες επιμόρφωσης. Να κοιτάξουμε επίσης και το θέμα των ε, χρηματοδοτικών μηχανισμών. Μήπως θα μπορούσε να υπάρξει και μια ανανέωση για να σχεδιαστεί ακόμα καλύτερα η δικαστική επιμόρφωση. Για όλους αυτούς τους λόγους λοιπόν, και λαμβάνοντα υπόψη τόσα σας είπα, που δεν είναι και τα μόνα, γιατί υπάρχουν και άλλα πράγματα που θα έπρεπε να, κοιμα... να κοιτάξουμε, ο Επίτροπό μου αποφάσισε να οργανώσει μια ευρεία διαβούλευση με όλου του ενδιαφερόμενου. Πολύ σύντομα θα αρχίσουμε με μια διαδικασία ανοιχτή διαβούλευσης τον Μάιο. Και εδώ πολλοί από εσά που βρίσκεστε σε αυτή την αίθουσα θα έχετε ήδη πάρει ερωτηματολόγια από εμά, έτσι ώστε η διαβούλευση αυτή να γίνει όσο γίνεται καλύτερα και να είναι όσο περισσότερο γίνεται ανταποκρινόμενη στις ανάγκες. Θα έχουμε και τον Νοέμβριο μεγάλη διάσκεψη προκειμένου να ακούσουμε τις ιδέες σας, τις στρατηγικές που προτείνετε, τις επιθυμίες σας και φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συνεισφέρει και η συνεισφορά του είναι κάτι παραπάνω από ευπρόσδεκτη. Βασιζόμαστε λοιπόν στη δικιά σας στήριξη, να μας βοηθήσετε να αναπτύξουμε μια καλή στρατηγική για την επιμόρφωση και πέρα από το 2020 για να προωθήσουμε την πολιτική μας επιμόρφωση σε θέματα δικαιοσύνης. Σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να είμαι η πρώτη που θα πάρω το λόγο σε αυτήν τη συνάντηση. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και προβλέπω στα σχόλιά σας. Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε για την οπτική αυτή από την Κομισιόν. Τώρα έχουμε περισσότερους βουλευτές που έχουν καταφτάσει. Σας ευχαριστώ γι' αυτό. Θέλω να υπογραμμίσω κάποια πράγματα σχέση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που το αναφέρατε. Καταρχήν και η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών έχουν δεσμευτεί σε αυτό το φιλόδοξο στόχο ε, της ε, κατάρτισης ε, των ασκούντων νομικά επαγγέλματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να φτάσουμε στους αριθμούς αυτούς ως το 2020. Εσείς αναφερθήκατε στο να στοχεύσουμε συγκεκριμένες χώρες και ε, τομείς ε, και χαίρομαι που βλέπω εδώ την τρεις ε, βουλευτές να είναι εδώ, είναι μέλη της Επιτροπής Λίμπε και τα μέλη της Επιτροπής Λίμπε και τα μέλη της Επιτροπής Γιούρι θέλουν να διατηρήσουν τη σχέση με τους συναδέλφους εδώ για να συμβεί κάτι τέτοιο και θέλουμε ποιοτική δράση, όχι μόνο ποσοτική. Τώρα, μπορούμε να περάσουμε στην ομιλία των εμπειρογνωμόνων. Θέλω να καλωσορίσω την Τατιάνα Τερμάτσιτς, η οποία είναι επικεφαλής του Τμήματος Εθνικής Εφαρμογής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ε, την κυρία Παστρέλα που είναι επικεφαλής της Μονάδας HELP. Ε, ουσιαστικά το HELP ε, σημαίνει εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα για τους ασκούντες νομικά επαγγέλματα και είναι η πλατφόρμα του Συμβουλίου της Ευρώπης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δικαστές, εισαγγελείς και δικηγόρους. Καταρχήν θα ακούσουμε την Τατιάνα. Θα ακολουθήσει η κυρία Παστράνα, η οποία είναι επικεφαλής ε, της μονάδας HELP για το Συμβουλίο της Ευρώπης. Παρακαλώ, Τατιάνα. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας ε, κυρίες και κύριοι. Καταρχήν ε, θέλω να ευχαριστήσω τα μέλη της Επιτροπής Γιούρη και της Επιτροπής Λίμπε, το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο που μας ε, κάλεσαν εδώ να παρουσιάσουμε το πρόγραμμα HELP του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τα τελευταία χρόνια έγινε το HELP η κύρια δύναμη σε ό,τι αφορά την νομική κατάρτιση ε, σε ό,τι αφορά τα θεμελιώδη δικαιώματα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Καλύπτεται 47 μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης. Ε, φυσικά εδώ ανήκουν και τα ευρωπαϊκά κράτη-μέλη. Έχουμε τρεις ε, συνιστώσεις στο HELP. Πρόκειται για ένα δίκτυο σχολών για τους δικαστές και τους εισαγγελείς και τους δικηγορικούς συλλόγους στα 47 κράτη-μέλη και φυσικά ε, έχουμε και εταίρου όπως είναι το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάρτιση Δικαστών και το Συμβούλιο Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, δεύτερον, ε, είναι μια πλατφόρμα με δωρεάν επιγραμμικά μαθήματα όπου εκεί έχουμε γνώση, αξίες και προσόντα δεξιότητε και τρίτον μεθοδολογία. Το HELP ουσιαστικά δεν υποκαθιστά το ρόλο των Εθνικών Ιδρυμάτων Κατάρτισης, αλλά τους δίνει συγκεκριμένα εργαλεία κατάρτισης που έχουν αναπτυχθεί από εμπειρογνώμονες του Συμβουλίου της Ευρώπης ε, που ουσιαστικά βασίζονται στο δίκαιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η πρωτότυπη προσέγγιση είναι ότι τα εργαλεία HELP θα ε, ουσιαστικά συγχωνεύσουν την εθνική προοπτική με την προοπτική, με την οπτική του Συμβουλίου της Ευρώπης έτσι ώστε τα ευρωπαϊκά πρότυπα να μην τα βλέπουμε ως ε, μία ξένη πηγή δικαίου. Έτσι λοιπόν, ε, πώς γεννήθηκε το χέλπ; είχαμε ε, ουσιαστικά ε, μία επιτροπή για την κατάρτιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα για τους ε, ασκούντες νομικά επαγγέλματα και τους φοιτητέ. Τότε χρειάστηκε ουσιαστικά να μεταρρυθμίσουμε το δικαστήριο για να μην καταρρεύσει, αλλά και να βελτιώσουμε την εφαρμογή της σύμβασης σε εθνικό επίπεδο. Και ένας από τους τρόπους να το κάνουμε αυτό ήταν φυσικά η νομική κατάρτιση, η οποία θεωρείται ένα διάκοπτο, ένα διάλειπο ταξίδι από το πανεπιστήμιο μέχρι την επαγγελματική στεδιοδρομία. Ο στόχο του HELP είναι να διασφαλίσει ότι η κατάρτιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα θα είναι υψηλή ποιότητα σε όλο τον ευρωπαϊκό χώρο και επίση ότι θα σέβεται θα απαντά σε όλε τι ειδικέ ανάγκε κάθε κατηγορία επαγγελματιών, δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων. Τα μαθήματα του HELP καλύπτουν όχι μόνο την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, αλλά και άλλες συμβάσεις του Συμβουλίου της Ευρώπης, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα και από το 2015 την ε, χάρτα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θεμελιώδη δικαιώματα, καθώς και την ομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Επίσης συνεργαζόμαστε με το ΦΡΑ, τον Οργανισμό για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και φυσικά έχουμε αναπτύξει ε, ένα μάθημα για την προστασία των δεδομένων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά είναι ο σύμμαχός μας, είναι ο φυσικός μας σύμμαχος και το 2015 το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέλαβε το μεγαλύτερο project κατάρτισης που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θεμελιώδη δικαιώματα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ονομάστηκε HELP στους 28. Και αυτή ήταν η συνεισφορά του HELP και του Συμβουλίου της Ευρώπης για να πετύχουμε αυτό το στόχο τον οποίο ακούσαμε νωρίτερα. Χωρίς την Ευρωπαϊκή Ένωση θα είχαμε περιορισμένο αντίκτυπο. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι πρέπει να ενδυναμώσουμε την εταιρική σχέση με το Συμβούλιο της Ευρώπης για να ωφελήσει περισσότερο το help της ευρωπαϊκές χώρες αλλά και τους νομικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να ε, καταστήσουμε το επάγγελμά τους πιο βιώσιμο πολυετός. Αυτό θα συνεισφέρει στο να οικοδομήσουμε την ευρωπαϊκή δικαστική κουλτούρα και θα ενισχύσουμε την ε, εμπιστοσύνη μεταξύ των νομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά θα προωθήσουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα σας ε, δώσω μία σύντομη εισαγωγή για το μάθημα για την προστασία των δεδομένων που είναι λιγότερο από δύο λεπτά. Πρέπει να ξεκινήσει τώρα το βίντεο. Hello, I'm Frank. A woman showed up in my law firm one afternoon with an unusual case. Γεια σα, είμαι ο Φρανκ. Πριν από λίγο καιρό ήρθε μια κυρία στο δικηγορικό μου γραφείο για μια συνήθιστη υπόθεση. Χρειάζομαι τη βοήθειά σα, είπε και εξήγησε ότι την απόλυσε το αφεντικό τη γιατί απίστωσε ότι είχε χρησιμοποιήσει το επαγγελματικό τη λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για προσωπικά mail και ότι επισκέφθηκε κοινωνικά δίκαια μέσα στο ωράριο εργασία τη. Και με ρώτησε, λοιπόν, μπορεί να με απολύσει σύμφωνα με τον νόμο το αφεντικό μου. Λίγο αργότερα μπήκα στη ιστοσελίδα του βακάλι μου για να παραγγείλω. Μόλι μπήκα, αμέσω μου προτάθηκαν κάποια προϊόντα πριν καν αρχίσω να διαλέγω. Μα πώ ξέρουν ότι εγώ χρειάζομαι γάλα ή πώ ξέρουν ποιο είναι το αγαπημένο μου κρασί. Αν είστε λοιπόν δικηγόρο, εισαγγελέα ή δικαστή και έχετε συχνά υποθέσει αντιμετωπίσετε προστασία δεδομένου ιδιωτικού βίου, τότε αυτό το ηλεκτρονικό μάθημα μπορεί να σα βοηθήσει. Έχει δημιουργηθεί με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο τη Ευρώπη. Είναι το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Κατάρτιση Νομικών σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, το γνωστό μα HELP. Θα σα βοηθήσει να καταλάβετε καλύτερα τι δυσκολίε που έχουν να κάνουν με την προστασία του ιδιωτικού βίου και με την προστασία των δεδομένων και θα μπορέσετε έτσι πιο εύκολα να προστατεύσετε τα δικαιώματα αυτά. Αποτελείται από 10 τμήματα. Τα πρώτα τρία είναι βασικέ γνώσει σχετικά με το δικαίωμα στον ιδιωτικό βίο και την προστασία των δεδομένων. Θα μάθετε τα νομικά μέσα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που απορρέουν είτε από το Συμβούλιο τη Ευρώπη είτε από την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιο είναι ο ρόλο των θεσμών και ποιε είναι οι βασικέ έννοιε, κανόνε και αρχέ. Τα επόμενα πέντε τμήματα παρουσιάζουν διάφορε προβληματικέ περιπτώσει που έχουν να κάνουν με την υγεία, τα μέσα ενημέρωση, τι νέε τεχνολογίε, τι ηλεκτρονικέ επικοινωνίε και παρακολουθούν παρακολούθηση στου χώρου εργασία. Και τα τελευταία δύο μαθήματα έχουν να κάνουν με τη συμμόρφωση με του κανόνε προστασία δεδομένων και ιδιωτικού βίου. Μην ξεχνάτε, το μάθημα έχει σχεδιαστεί για να ανταποκρίνεται στι δικέτερε ανάγκε των νομικών. Περιλαμβάνει πολλά πρακτικά παραδείγματα για να εξοικειωθείτε με τι τρέχουσε εξελίξει στην δικαιοσύνη. Ολοκληρώνοντα επιτυχώ το μάθημα, λαμβάνετε και επιστοποιητικό help. Για περισσότερε πληροφορίε επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μα. Καλή τύχη! Good afternoon. Καλησπέρα σας. Τώρα είναι η σειρά μου. Λέγομαι Βουκαστράνα και είμαι εδώ σήμερα για να μιλήσω για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ε, κατάρτιση των δικαστικών. Ε, πάντοτε ξεκινάμε με μια ιστορία στα μαθήματά μας και εγώ θα ξεκινήσω με τη δική μου. Για 13 χρόνια εργαζόμουν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε τόπους όπως οι Φιλιππίνες, η Νικαράγουα, η Γεωργία και κατόπιν ε, ε, έφυγα από την Κομισιόν και έρχισα να δουλεύω για το Συμβουλίο της Ευρώπης. Τώρα εργάζομαι για το Συμβουλίο της Ευρώπης και μπορώ να, ακολουθήσω τα δύο πάθη μου, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το ευρωπαϊκό έργο. Και νομίζω ότι τα ίδια πάθη σας καθοδηγούν και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Έτσι λοιπόν, το σχέδιο σήμερα είναι να σας παρουσιάσω τι είναι το HELP. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ίδρυσε το HELP στις 28 χώρες. Γιατί τώρα, επίση, πρέπει να σα παρουσιάσω, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το Συμβούλιο τη Ευρώπη πρέπει να ενώσουν τι δυνάμει του για να υπερασπίσουν καλύτερα τα ανθρώπινα δικαιώματα αν έχουμε χρόνο, θα σα ε, έλεγα να δούμε και τι γίνεται και με τα εργατικά δικαιώματα. Ουσιαστικά, εδώ ε, έχουμε προσθέμενη αξία του HELP. Ε, εμείς παρακολουθούμε τα απορίσματα και ενεργοποιούμε τους καλύτερους συναδέλφους και έτσι λοιπόν εμείς στο HELP είμαστε στην καλύτερη θέση για να αναπτύξουμε τα καλύτερα μαθήματα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι λοιπόν... Εδώ πρόκειται για μια οπτική υπενθύμηση σε σχέση με όσα είπε η Τατιάνα. Το δίκτυο HELP που συμπεριλαμβάνει ε, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Κατάστασης Δικαστών ε, και το Συμβούλιο Δικηγορικών ε, Συλλόγων. Με το EJTN επικεντρωνόμαστε στα ανθρώπινα δικαιώματα αλλά καλύπτουμε και τους δικηγόρους. Έχουμε την πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης με μαθήματα δωρεάν που είναι διαθέσιμα για όλους. Και έχουμε την ε, μεθοδολογία κατάρτισης για τα ανθρώπινα δικαιώματα και φυσικά έχουμε έτσι υψηλό επίπεδο κατάρτισης. Προσπαθούμε λοιπόν να υιοθετήσουμε αυτό το περιφερειακό σχέδιο. Εργαζόμαστε μερικές φορές σε δύσκολες περιφέρειες όπως τα Δυτικά Βαλκάνια ή χώρες όπως η Ρωσία και για την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Χάρη στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούσαμε να εφαρμόσουμε το πρόγραμμα για τα 28 κράτη-μέλη και μπορούσαμε να παράσχουμε στους επαγγελματίες γνώση και ε, για να μπορούν να εφαρμόσουν την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων ε, Δικαιωμάτων, ε, την Ευρωπαϊκή Κοινωνική Χάρτα και όλη τη σχετική νομοθεσία. Εμείς αναπτύξαμε μαθήματα που ουσιαστικά συγχωνεύουν το σύστημα της Συμβουλίου της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουμε συμπεριλάβει την ομολογία και του Στρασβούργου και του Λουξεμβούργου. Έτσι λοιπόν, κατά πολέμηση, κατά του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, της ομοφοβίας και την τρανσφοβία. Ε, ξέρετε ότι έχουμε ρατσισμό και ξενοφοβία λόγω της υψηλής ζωής προσφύγων. Επίσης είχαμε ε, ένα μάθημα για την προστασία των δεδομένων, ε, εργατικά δικαιώματα, εργασιακά δικαιώματα. Πρέπει να υπερασπίσουμε τα εργασιακά δικαιώματα σε καιρούς κρίσης και ε, ουσιαστικά πρόθετας και την πλήρη επασχόληση, τα δικαιώματα για την ακαιρεότητα του προσώπου, επικεντρώμαστε στη βιοεθική. Πρόκειται για πάρα πολύ ευαίσθητα θέματα, όπως το χάρη τον, τερματικό της, ε, τερματισμό της ζωής ή ε, της ε, μητέρες. Και επίσης ε, έχουμε επικεντρωθεί και σε μια κοινή δήλωση Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πέρα από αυτά τα μαθήματα έχουμε και ένα κατάλογο για τα θεμελιώδη δικαιώματα και έχουμε εδώ εναλλακτικά μέτρα της κράτησης, δικαιώματα ιδιοκτησίας, ε, ε, ε των αιτιολόγηση των δικαστικών ε, αποφάσεων. Βλέπετε εδώ διάφορα θέματα, τα έχετε στη διάθεσή σας. ήθελα να σας δείξω ποιος είναι ο αντίκτυπος ε, των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Πρόκειται για χρήματα του Ευρωπαίου Φορολογουμένου και τα έχουμε χρησιμοποιήσει σωστά. Ξεκινήσαμε 25 μαθήματα σε 16 κράτη-μέλη ε, και ε, ουσιαστικά απευθυνθήκαμε σε 750 δικαστικούς και είχαμε και ευρύτερο κρατήριο. Όμως χρειαζόμαστε περισσότερα μαθήματα, χρειαζόμαστε περισσότερες προτεραιότητες και πρέπει να καλύψουμε όλες τις χώρες. Βλέπετε λοιπόν εδώ τον αντίκτυπο της χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τριπλασιάσαμε την ε, τακτική δουλειά του Συμβουλίου της Ευρώπης στις ευρωπαϊκές χώρες και μπορούμε να δεσμεύσουμε, να εμπλέξουμε και πάρα πολλές εθνικές ενώσεις. Ελπίζουμε να έχουμε την υποστήριξή σας σε αυτά. Και τώρα να σας δείξω αυτό το γράφημα που είναι πολύ γλαφυρό. Βλέπουμε μια τεράστια αύξηση των χρηστών της πλατφόρμας μας. Είχαμε 18.000 τριπλασιάσαμε τον αριθμό των χρηστών το 2016. Το 2016 είχαμε τέσσερις φορές περισσότερους χρήστες από το 2014 και Κάτι ακόμη πιο εντυπωσιακό, μόνο το πρώτο τρίμηνο του 2017 σχεδόν είχαμε τον ίδιο αριθμό νέων χρηστών με το 2016. 6.000 άτομα δηλαδή που άνοιξαν λογαριασμό στην πλατφόρμα μας. Επομένως, φτάνω προς το τέλος. Θέλω να ζητήσω την υποστήριξή σας ε, για να έχουμε νομοθεσία και πόρους για να υποστηρίξουμε την κατάρτιση δικαστικών στην Ευρώπη. Έχουμε υψηλέ ε, προσδοκίε, βραχυπρόθεσμα. Έχουμε υποβάλει δύο προτάσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμω έχουμε και ψηλότερε προσδοκίε, ε, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Γιατί, αν θέλουμε σοβαρά να αντιμετωπίσουμε τις πολυάριθμες προκλήσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα, χρειαζόμαστε πόρους και πρέπει να το παραδεκτούμε, γιατί το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει πάρα πολύ περιορισμένους πόρους. Σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο προπολογισμό του Συμβουλίου της Ευρώπης είναι 0,29% του συνολικού ενωσιακού προπολογισμού. και τα κράτη-μέλη το ξέρουν αυτό πάρα πολύ καλά αλλά δεν είναι πρόθυμα να δώσουν χρήματα σε εμά, γιατί μας θεωρούν ε, ε, ουσιαστικά ότι ασκούμε πάρα πολύ δρυμία κριτική όταν ε, πρόκειται για ανθρώπινα δικαιώματα. Αν ε, μπορούσαμε να θεωρήσουμε τη στρατηγική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση και ενώσουμε τις δυνάμεις μας, αν λάβουμε ένα εκατομμύριο ευρώ επιπλέον ετησίως θα τριπλασιάσουμε τον αντίκτυπό μας. Και γι' αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να συνεχίσουμε. Είπε η Αλεσάνδρα ότι τα χρήματα βοηθούν, αλλά και το help χρειάζεται βοήθεια. Έτσι λοιπόν θα συμβάλλουμε στο να βελτιώσουμε αυτή την κουλτούρα, την ευρωπαϊκή κουλτούρα των δικαστικών που χρειάζεται και να υποστηρίξουμε τις ευρωπαϊκές αξίες. Ευχαριστώ πολύ. Μάλιστα. Ευχαριστώ για το έτοιμά σας. Και τώρα θα περάσουμε στην Βαλερή Σαγκάντ. Ε, θα συνεχίσω στα γαλλικά. Ευχαριστώ πολύ για τόσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Πολύ ενδιαφέροντα και είναι κρίμα πραγματικά που δεν υπάρχουν εδώ πέρα περισσότεροι παρόντες. Αλλά είμαι πεπισμένη ότι η συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης Ευρωπαϊκή Ένωση, Συμβούλιο της Ευρώπη δηλαδή, είναι κάτι από το οποίο έχουν αποφεληθούν όλοι ασχολούνται με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Τώρα, οι επιρρογνώμονε, παρακαλώ, του Ευρωπαϊκού Δικτύου επιμόρφωση σε θέματα δικαιοσύνη που είναι ειδική σε θέματα βέλτιστων πρακτικών στην επιμόρφωση αυτή και θα μας ενημερώσουν για τις ανταλλαγέ που γίνονται στο δικαστικό τομέα. Έχουμε δύο μέλη από δύο εθνικά και σχολές δικαστών, Γαλλίας και Βελγίου και τον ε, Μέτρε Σράντερ, ο οποίος συμμετείχε πρόσφατα ως πρόεδρος ε, ενός εφετείου σε κάτι στην ε, Γερμανία. Είναι όλοι στην καλύτερη δυνατόν θέση για να μας ενημερώσουν για τις ανταλλαγές αυτές. Οπότε, από την ε, Γαλλική Σχολή Δικαστών πρώτα και μετά από το Βέλγιο. Η κυρία Σαγκάντ πρώτα λοιπόν και μετά ο κύριος Φαν Ράντσπεκ από το Βέλγιο. Θα ξεκινήσετε εσείς κυρία Σαγκάντ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, αυτό το δίκτυο δικαστικής κατάρτισης δημιουργήθηκε το 2000 και συμμετέχουν εκεί όλα τα Ινστιτούτα, όλες οι σχολές που ε, εκπαιδεύουν δικαστές και νομικούς στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπατε, χρηματοδοτείται κυρίως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και υπάρχουν και καμιά κοσαριά άνθρωποι εδώ στις Βρυξέλλες που συμμετέχουν επίσης βάσει της βελγικής δικαιοσύνης. Αλλά πάνω απ' όλα βασιζόμαστε στις ίδιες τις σχολές εκπαίδευσης και στις δυνατότητες που έχουν να αναλύσουν και τις ανάγκες των συναδέρφου τους σε θέματα επιμόρφωσης και να φροντίσουν να δώσουν και να προσφέρουν την εκπαίδευση και κατάρτιση ακριβώς που χρειάζεται. Έχουμε εμπειρία 10 ετών. Πολλαπλησιάστηκαν επί 10 οι ημέρες επιμόρφωσης. Είναι 30.000 περίπου που προσφέρουμε σήμερα και πάνω από 5.000 δικαστές και εισαγγελείς συμμετέχουν. Στόχος μας είναι να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή δικαστική παράδοση με γνώση βέβαια και του ευρωπαϊκού δικαίου, την ομολογία του ευρωπαϊκού δικαστηρίου, ε, συγκεκριμένα πώς μπορούν οι προσανατολισμοί αυτοί να τεθούν στην πράξη και να υπάρχει και συνεργασία μεταξύ μας. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν ανταλλαγές και θα τα ακούσετε αυτά και αργότερα από τους συναδέλφους. Πολλές είναι οι δραστηριότητές μας και έχουν να κάνουν με σεμινάρια επιμόρφωσης πρώτα απ' όλα τρεις, τέσσερις και πέντε μέρες μερικές φορές, ανάλογα με τα θέματα. Έχουμε και ηλεκτρονική επιμόρφωση. Υπάρχουν κάποια μαθήματα τώρα τέτοιες ηλεκτρονικής επιμόρφωσης, ώστε οι συμβολογράφοι και οι δικαστές, σε συνεργασία με τους συμβολογράφους ακριβώς, να παρακολουθούν τέτοια ηλεκτρονική επιμόρφωση για θέματα, ας πούμε, κληρονομικά. Προσπαθούμε να ανταποκριθούμε λοιπόν στις ανάγκες των Ευρωπαίων πολιτών είναι επίσης μια δραστηριότητα και αυτή οι ανταλλαγές. Όλες αυτές οι δραστηριότητες μας οδήγησαν στο να εντοπίσουμε κάποιες αρχές που θέλω να σας παρουσιάσω, όχι τόσο επειδή πρόκειται για αρχές, αλλά για να σας εξηγήσω πόσο μεγάλη σημασία έχει ο ρεαλισμός στο δίκτυο αυτό. Το δίκτυο λοιπόν έχει καταλήξει σε νέα θεμελιώδεις αρχές σε θέματα δικαστικής επιμόρφωσης. Το πρώτο έχει να κάνει με το ότι η επιμόρφωση αυτή πρέπει να είναι και επαγγελματικού χαρακτήρα αλλά και πολυτομιακή. Εμείς επιμένουμε στο πρακτικό χαρακτήρα της επιμόρφωσης, γιατί δεν πρόκειται για ακαδημαϊκή μόρφωση. Εμείς θεωρούμε ότι το δίκαιο, γνώση δηλαδή του δικαίου υπάρχει ήδη, ότι γνωρίζουν το ευρωπαϊκό δίκαιο οι άνθρωποι αυτοί. Αυτό όμως που θέλουμε είναι να επικεντρωθούμε σε πρακτικά ζητήματα που έχουν να επιλύσουν οι άνθρωποι αυτοί στην καθημερινή τους επαγγελματική ζωή. Η επιμόρφωση αυτή πρέπει να είναι επίσης υποχρεωτική. Πρέπει να υπάρχει αυτό το δικαίωμα στην επιμόρφωση. Όλα αυτά είναι αναγκαία. Να υπάρχει φυσικά και ανεξαρτησία στη δικαιοσύνη εννοείται, το δικαίωμα στην κατάρτιση. Ε, κάτι άλλο στο οποίο επιμένουμε πολύ και μας βοηθάει το δίκαιο είναι πώς θα επιμορφώσουμε τους δικούς μας τους δασκάλους, αυτούς που προσφέρουν στη συνέχεια επιμόρφωση. Είναι δικαστές, είναι εισαγγελείς, είναι δικηγόροι, συμβολιογράφοι, είναι προσωπικό επίσης των δικαστηρίων και όλοι αυτοί είναι άνθρωποι που στην πράξη ασχολούνται με αυτά τα θέματα. Πρέπει όμως να γνωρίζουν και λίγο από παιδαγωγική. Πόσο δηλαδή να διδάξουν με τη συμμετοχή όλων, με προσωμιώσεις και να υπάρχουν και ανταλλαγές πληροφοριών για αυτού του είδους την εκπαίδευση, για αυτού του είδους τα εργαστήρια δηλαδή, στα οποία εκπαιδεύονται οι επιμορφωτές. Εννοείται ότι χρειάζονται επαρκή σπόρη για να γίνει αυτό και χρειάζεται και η στήριξη των ανώτατων δικαστικών αρχών. Κάτι το οποίο το έχουμε καταφέρει στις περισσότερες από τις χώρες μας, αλλά κάθε φορά πρέπει να δίνουμε αγώνα για να το πετύχουμε. Εντοπίσαμε επίσης και κάποιες προκλήσεις για το μέλλον. Πέρα από το ζήτημα της γλώσσας, πρέπει να αναπτύξουμε επιμόρφωση για όλους τους δικαστές και τους εισαγγελείς και όχι μόνο για αυτούς που προέρχονται από μια ευρωπαϊκή παράδοση. Αυτή είναι μια δυσκολία που αντιμετωπίζουμε και προσπαθούμε να προχωρήσουμε και πάνω σε αυτό. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Στα Ολλανδικά θα προχωρήσω εγώ. Στόχος μας είναι τώρα να προχωρήσουμε λίγο περισσότερο στο θέμα της ανταλλαγής και στο ποιο ρόλο το δίκτυο αυτό μπορεί να παίξει στην οργάνωση τέτοιων ανταλλαγών με τρίτους. Αυτό που είναι σημαντικό εδώ και το λέμε και το ξαναλέμε είναι το δίκτυο αυτό επιμόρφωσης για την Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη. Είναι ένα δίκτυο που συμμετέχουν σχολές και όργανα που είναι αρμόδια για την κατάρτιση των δικαστών και ορισμένοι μάλιστα είναι αρμόδιοι και για, άλλες, ε, για άλλους κλάδους, αλλά εμείς κυρίως ε, με τους δικαστές ασχολούμαστε. Το δίκτυο αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ εντατική ανταλλαγή πληροφοριών και επίσης αποτελεί την κατεξοχήν πλατφόρμα το δίκτυο αυτό για να προχωρούν και προγράμματα ανταλλαγής πληροφοριών. Το είδατε και στο γράφημα που πριν σας έδειξε η Βαλερή ότι τα προγράμματα ανταλλαγή πρέπει να είναι προγράμματα που να αποτελούν ό,τι πιο εμβληματικό για το δίκτυό μας. Ήδη από το 2005 ξεκινήσαμε, τότε είμαστε κάπου 170 συμμετέχοντας μόνο, ενώ σήμερα είναι 2.200 οι συμμετέχοντες που έχουν τη δυνατότητα δηλαδή να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους ανταλλαγές. Μέσα σε 10 χρόνια, 12 χρόνια δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι η πρόοδος είναι τεράστια. Με τον ένα με τον άλλο τρόπο, λοιπόν, συμμετέχουν όλο και περισσότεροι και ενημερώνονται για το ευρωπαϊκό δίκαιο Πρόκειται τώρα και για δικαστές και εισαγγελείς, νομικούς από μια χώρα που βρίσκονται με συναδέλφους τους από μια άλλη χώρα. Υπάρχει ανταλλαγή επίσης προσώπων που βοηθάει σε πλούτο εμπειριών και σε ενημέρωση όσον αφορά τις βέλτιστες πρακτικές. Τώρα τα προγράμματα μας ανταλλαγών. Πώς έχουν. Έχουμε τρία είδη ανταλλαγέ. Έχουμε τι βραχυπρόθεμε ανταλλαγέ, δηλαδή πρόκειται για ανταλλαγέ που κρατάνε μία-δύο εβδομαδε και οι δικαστέ μιας χώρας πάνε σε μια άλλη χώρα για να ενημερωθούν και να καταλάβουν καλύτερα πώς λειτουργεί το δικαστικό σύστημα στην άλλη χώρα. Η δεύτερη περίπτωση είναι study visits, αλλά και μακροχρόνια κατάρτιση. Study visits είναι επισκέψεις που γίνονται ε, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, λοιπόν, στη Eurojust ή αλλού και υπάρχει δυνατότητα όμως να παραμείνουν οι άνθρωποι αυτοί και μακροχρόνια σε τέτοια όργανα, τρεις μήνες έως και ένα χρόνο. Και η τρίτη περίπτωση είναι το πρόγραμμα Αγιάκος, που είναι ένα πρόγραμμα ανταλλαγών που επικεντρώνεται σε νέους που μπαίνουν στο δικαστικό σώμα ή στην επιμόρφωση των δικαστικών. Παρά την επιτυχία και παρά το γεγονός ότι ένα μεγάλο μέρος του δικαστικού σώματος έχει ευαισθητοποιηθεί ε, στο θέμα των ανταλλαγών, οι προκλήσεις παραμένουν. Το θέμα της γλώσσας είναι μια μεγάλη πρόκληση, γιατί δεν είναι εύκολο άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τόσο καλά μια ξένη γλώσσα να πηγαίνουν σε μια ξένη χώρα δεν θεωρούν ότι έχουν κίνητρο να το κάνουν. Είναι ένα θέμα το οποίο εμείς παρακολουθούμε, προσέχουμε και προσπαθούμε να το διορθώσουμε με μια καλύτερη οργάνωση. Υπάρχει το θέμα επίσης του χρόνου που έχουν στη διάθεσή τους, μάλλον που δεν έχουν οι δικαστές στη διάθεσή τους. Γιατί έχουν να διεκπαιρεώσουν ένα σωρό υποθέσεις και δεν είναι πάντα εύκολο να σταματήσουν τη δουλειά τους για να συμμετέχουν σε τέτοιου είδους ανταλλαγές. Γι' αυτό λοιπόν και θέλουμε να δουλεύουμε κατά περίπτωση. Λαμβάνουμε υπόψη μας τις ανάγκες σε περιβαλλοντικό δίκαιο, εργασιακό δίκαιο και άλλα. Και ένα, ένας ειδικός τομέας ανταλλαγών έχει να κάνει με αυτό για το οποίο θα σας μιλήσω ο συνάδελφος σε λίγο, που είναι η επικεφαλής των σωμάτων. Είπαμε, μας ενδιαφέρει η ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, αλλά συγχρόνως μας ενδιαφέρει και η μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση των ανθρώπων αυτών που είναι επικεφαλής σωμάτων, ώστε με τη σειρά τους να μπορέσουν να ευαισθητοποιήσουν περισσότερο τους εφισταμένους τους και να τους δημιουργήσουν περισσότερο ενθουσιασμό για τη δουλειά τους. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Σράντερ, ο οποίο έχει συμμετάσχει σε τέτοια προγράμματα ανταλλαγών. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ ε, κύριε Γάντσπεκ. Ε, θα ήθελα λοιπόν να σας ε, περιγράψω την δική μου εμπειρία στη Σλοβανία. Θα, στη Σλοβενία. Μία από τις δυσκολίες ήταν βέβαια η γλώσσα, διότι οι περισσότεροι δικαστές εργάζονται στη μετρική τους γλώσσα με αποτέλεσμα αυτό να αποτελεί μια δυσκολία διότι το γλωσσικό πρόβλημα δεν μπορεί να ξεπεριστεί. Επίσης το επίπεδο των αγγλικών μου ε, ήταν αρκετό ε, για να μπορέσω να συμμετάσχω. Επίσης ε, για πρώτη φορά γινόταν μια ανταλλαγή για προέδρους δικαστηρίων. Το γεγονός αυτό έλαβε χώρα στην Λιουμπιάν και συνεργαζόταν με το Υπουργείο Δικαιοσύνης της ε, Σλοβενίας. Ε, ε, ένας υπάλληλος λοιπόν του κέντρου αυτού μας εξήγησε το έργο του Ινστιτούτου, το οποίο είναι για παράδειγμα να προετοιμάζει για την αποδοχή, για την είσοδο στις εξετάσεις νομικής. Επίσης ένας δικαστής μας είπε ότι Στόχο τη Σλοβανία είναι να μειώσει τον αριθμό των ε, δικαστών, βελτιώνοντα την αποδοτικότητα του δικαστικού συστήματο. Επίση, συζητήσαμε ζητήματα ε, νομοθεσία και ήταν ξεκάθαρο ότι υπήρχαν μεγάλε προσδοκίε όσον αφορά την συμπεριφορά των δικαστικών, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε προσωπικό επίπεδο. Επισκέφθηκα ε, το ανώτατο εργατικό δικαστήριο και συζητήσαμε και εργατικά ζητήματα και συνειδητοποιήσαμε ότι οι συμβιβασμοί εκεί πέρα είναι πιο ασυνήθι σε σχέση με τη Γερμανία. Ε, επίσης, ε, στην Σλοβανία ε, ο δικαστής έχει το δικαίωμα να θέσει υποψηφίους και επίσης απαιτείται η έγκριση του Κοινοβουλίου. Ε, κάτι τέτοιο είναι πάρα πολύ ε, σύνηθες ε, στη χώρα. Οι δικαστές επίσης ε, υπόκεινται σε μια ετήσια εξέταση, εξέταση τα τρία πρώτα χρόνια εργασίας τους και ο στόχος αυτός ε, έχει ώστε ο πρόεδρος να λάβει στατιστικά δεδομένα με αποτέλεσμα να λάβει από το, το ανώτατο δικαστήριο μια άποψη και, και ακολουθείται παρόμοια διαδικασία και με τους διαδικαστές, για τους, τους ε, προανέφερα το γλωσσικό εμπόδιο. Πέρα από αυτό όμως δεν υπήρχαν άλλα εμπόδια τα οποία χρειάστηκε να ξεπεράσω. Ε, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της χώρας μου ε, παροτρύνει στη συμμετοχή σε τέτοια προγράμματα ενώ το Υπουργείο της Σλοβενίας καλωσόρισε τους ξένους δικαστές καθώς επίσης και τους εισαγγελείς η ανταλλαγή Έχει τη δυνατότητα να συγκρίνω τα δύο ε, δικαστικά συστήματα με διάφορους τρόπους. Ε, είχα υποδομητικές συζητήσεις με συνοδόλφους και για άλλη μια φορά συνειδητοποίησα ότι τα προβλήματα στη δικαιοσύνη στις ε, ευρωπαϊκές χώρες είναι κοινά σε ένα βαθμό. Θα πρέπει λοιπόν να αναζητήσουμε εξέφραση λύσεων και αυτό μπορεί να γίνει μέσω της κοινή κατανόησης των Ευρωπαίων δικαστών οι οποίοι θα μάθουν από τα ευρωπαϊκά δικαστικά, δικαστικά συστήματα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ για τη μαρτυρία σας και χωρίς χρονοτριβή θα δώσω το λόγο στον κύριο Πιέρ Τζοβάνι Τραβέσο, ο οποίος είναι πρόεδρος της Επιτροπής Κατάρτισης. Είστε και πρόεδρος του Συμβουλίου Δικηγορικών Συλλόγων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ που ήρθατε εδώ στις Βρυξέλλες και σας καλώ να μας παρουσιάσετε τις βελτίσεις πρακτικές ε, της δικής σας ένωσης. Να μας πείτε επίσης ε, και ποιες είναι οι πιο σημαντικές προκλήσεις για το μέλλον. και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ε, προέδρους των επιτροπών ε, για την ε, τιμή που μου δίνουν να με προσκαλέσουν σε αυτό το εργαστήριο στην καρδιά της Ευρώπης και μιλώντας εκ μέρους του, του Συμβουλίου Δικαστικών Συλλόγων της Ευρώπης είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε το τη δεκαετία του 1960 ε, και από την δημιουργία της ε, βρίσκεται στο επίκεντρο ε, της βελτίωσης της χρήσης του δικαίου στην Ευρώπη και της χρήσης νόμων πάνω στους οποίους βασίζεται η Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και το κράτος δικαίου. Συμμετέχουν σε αυτό 45 χώρες από την, από την Ευρωπαϊκή Οικονομική Ζώνη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, ενώ ε, έχουμε 32 πλήρη ε, μέλη και 10 χώρες παρατηρητές. Και συμμετέχουν πάνω από ένα εκατομμύριο Ευρωπαίοι δικηγόροι αυτό ε, έρχεται ύστερα από την πρόταση που έγινε στην αρχή του ε, εργαστηρίου να ακούσουμε όχι μόνο τις απόψεις των πλήρων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που είναι σε αυτούς τους συλλόγους αλλά να έχουμε και ένα ευρύτερο σενάριο και για τους παρατηρητές και τις συνδεδεμένε χώρες. Υποστηρίζουμε ε, λοιπόν τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δημιουργήσει μια δικαστική κουλτούρα σε έναν τομέα ε, κοινών αξιών και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Η αυξανόμενη ελεύθερη κυκλοφορία ανθρώπων και επιχειρήσεων στην νέα αγορά της Ευρώπης έχει δημιουργήσει την ανάγκη δικηγόρων οι οποίοι θα γνωρίζουν τα νομικά συστήματα των γειτονικών τους χωρών. Και την ε, βελτίωση του επαγγέλματό τους. Επίσης, η επιρροή της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας ε, σε έναν αυξανόμενο τομέα, ε, σε αυξανόμενο αριθμό τομέων σημαίνει ότι οι δικηγόροι θα πρέπει να έχουν μια καλή κατανόηση του πρωτογενούς και δευτερογενούς νομοθεσίας καθώς επίσης και να έχουν τα εργαλεία ώστε να εφαρμόσουν ορθά την νομοθεσία. Το CCB υποστήριζε πάντοτε την, ε, ε, α, την βέλτιστη εκπαίδευση των ε, νομικών και την κατανόηση των νομικών συστημάτων της Ευρώπης. Για παράδειγμα, ένα από τα έγγραφα του CCB που εκδόθηκαν το 2007 ήταν μια πρόταση για την εκπαίδευση των αποτελεσμάτων δικών για δικηγόρους όπου τονίζεται ότι ο ο κάθε δικηγόρος εφαρμόζει την ε, καθημερινή του ε, δουλειά και ακολουθείται ένα πρότυπο πάνω στον οποίο γίνεται ε, το έργο διότι θα πρέπει να θυμόμαστε ότι το CCB αυτό καθ' αυτό δεν είναι ένα σώμα εκπαίδευσης. Έχουμε μια εκπαιδευτική επιτροπή στο εσωτερικό του CCB όμως αυτό, αυτή η επιτροπή δίνει προτάσεις όσον αφορά την εκπαίδευση δικηγόρων τόσο, τόσο στην αρχή της της εκπαίδευσης όσο και στη συνεχιζόμενη φάση. Έχουμε 36 μέλη από 19 χώρες και ε, ε, συναντώνται 5 φορές το χρόνο. Και οι δικηγόροι είναι ε, πάντοτε ευγνώμονες που έρχονται σε επαφή με ευρωπαϊκούς θεσμούς και επιθυμούν όσο τη δυνατόν περισσότερη υποστήριξη σε εκπαιδευτικά ζητήματα η εκπαιδευτική δομή για δικηγόρους ε, διαφέρει από χώρα σε χώρα. Ε, η ρύθμιση για την εισαγωγή στο επάγγελμα αλλά και η εγγραφή των δικηγόρων είναι μία από τις βασικές λειτουργίες ε, των ε, συλλόγων δικηγόρων της Ευρώπης, των δικηγορικών συλλόγων. Θέλουμε να διασφαλίσουμε τα ανώτατα επίπεδα εκπαίδευσης. Όλες οι χώρες ε, έχουν μια σειρά προτύπων και κανόνων σχετικά με το ποιος μπορεί να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο επάγγελμα. Στις περισσότερες χώρες απαιτείται να κατέχετε ένα μεταπτυχιακό ε, σε, στη νομική από ευρωπαϊκές χώρες να υπάρχει ε, πρακτική εμπειρία ή να έχει γίνει κάποια άσκηση καθώς επίσης και να ε, περάσει τελικές εξετάσεις. Όλα αυτά συνδέονται και με το ερώτημα σχετικά με το ότι κάθε χώρα έχει τις ιδιαιτερότητές της, τις παραδόσεις της και ε, προσπαθούμε να βρούμε μια ισορροπία ε, μεταξύ μεταξύ των προτύπων ε, που απαιτώνται για να γίνει κάποιος μέλος του δικηγορικού συλλόγου. Η ε, συνεχιζόμενη κατάρτιση, η διαβίου κατάρτιση είναι αναγκαία σε 17 χώρε όπω είναι η Εστονία, η Δανία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Γερμανία, η Ιρλανδία, η Ιταλία, η Λετωνία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Πολωνία, η Ρουμανία, η Σουηδία, οι ε, κατοχώρε, το Ηνωμένο Βασίλειο, και συγκεκριμένα ε, στην, ε, και στην Αγγλία, ε, στην Ουαλία, στη Σκωτία και στη Βόρεια Ιρλανδία. Έχουμε επίσης την Ελβετία και την Νορβηγία η ε, αγορά εκπαίδευση είναι ανοιχτή, με άλλα λόγια δηλαδή. Οι δικηγόροι μπορούν να αλλάξουν από μια σειρά δραστηριοτήτων διαβίου εκπαίδευση που προσφέρονται από δικηγορικούς συλλόγους, ε, πιστοποιημένους παρόχους εκπαίδευσης, ε, καθώς επίσης και παρόχους της ελεύθερης αγοράς. Ε, αναλυτικές λεπτομέρειες ε, σχετικά με ε, την υποχρέωση για την εκπαίδευση για κάθε χώρα βρίσκεται, είναι διαθέσιμη στα, στους εθνικούς πληροφοριακούς καταλόγους που έχουν κατατεθεί σχετικά με την κατάσταση της εκπαίδευσης δικηγόρων στην Ευρώπη από το 2014. δύο βασικά προγράμματα εκπαίδευσης ε, τα οποία ε, οργανώθηκαν από το CCB χάρη ε, στην ευρωπαϊκή χρηματοδότηση είναι η έρευνα η οποία προαναφέρθηκε σχετικά με την κατάσταση εκπαίδευσης δικηγόρων στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και ολοκληρώθηκε με την, με την έκδοση μιας μελέτης το 2014 η μελέτη λοιπόν προτείνει το νομικό επάγγελμα να, να συμπεριλάβει ε, ένα ε, πρόγραμμα σπουδών το οποίο θα περιλαμβάνει και το ευρωπαϊκό δίκαιο και θα περιλαμβάνει δραστηριότητες εκτός, εκτός συνόρων με αποτέλεσμα να γίνει ε, πιο στοχευμένο στην πρακτική άσκηση και να υπάρχει πρόσβαση στην εκπαίδευση και να υπάρχουν περισσότερες εκπαιδευτικές συναντήσεις και αλλαγές. Επίσης η μελέτη περιλαμβάνει πληροφορίες για τα εκπαιδευτικά εκπαιδευτικά συστήματα για τους δικηγόρους ανά χώρα, τα οποία καλά, καλύπτουν τόσο την αρχική όσο και τη συνεχιζόμενη τη διαβίω κατάρτιση. Το Νοέμβριο του 2014 τώρα το CCB οθέτησε στις ε, Βρυξέλλες στην Ολομέλεια του ένα σχέδιο δράσης ε, για να προωθήσει τις συγκεκριμένες προτάσεις Σήμερα λοιπόν το CCB έχει εργαστεί πάνω σε μια κοινή αναγνώριση της διαβίους, ε, διαβίου εκπαίδευσης δικηγόρων, στο οποίο ε, θα αναφερθώ εντός ολίγης, εν ολίγης. Το ε, Ίδρυμα Ευρωπαίων Δικηγόρων έχει ε, τον βασικό στόχο να εφαρμόσει ε, προγράμματα προστιθέμενης αξίας για δικηγόρους σε ζητήματα τα οποία σχετίζονται με πολιτικές ε, για δικαστές και ξεκίνησε ένα πόρταλ εκπαίδευσης το Σεπτέμβριο του 2014 το οποίο προσφέρει ορατότητα σε πρωτοβουλίες της Ευρώπης για την εκπαίδευση των νομικών. Το άλλο σημαντικό project το οποίο προωθήσαμε, το οποίο κάναμε είναι η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα Εκπαίδευσης για Δικηγόρους και ο στόχος αυτής της ε, πλατφόρμας είναι να καλύψει την έλλειψη προφόρησης σχετικά με τα ε, μαθήματα ε, πάνω στη νομική κατάρτιση και είμαι ιδιαίτερα περήφανος για το συγκεκριμένο project διότι είδα, διότι το παρακολούθησε από τα σπάργανά του στο εσωτερικό της Επιτροπής όπου είχαν βρεθεί ειδικοί από την Ιταλία, την ε, Γαλλία και τη Δανία και η όλη ιδέα χαιρετήθηκε από το CCB το οποίο υπέβαλε αίτηση για χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα λοιπόν εμείς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργαζόμαστε ε, για την συμπερίληψη της ε, πλατφόρμας ε, στο πόρταλ του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, το οποίο θα περιλαμβάνει έναν αναλυτικό κατάλογο μαθημάτων, καθώς επίσης και υλικό κατάρτισης. Οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθούν μαθήματα, τα οποία προσφέρονται σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ θα μπορούν να βλέπουν ε, τον τίτλο του ε, μαθήματος, σε ποια γλώσσα θα γίνεται, πού και πότε, ε, ποιο παρέχει. Οι πάροχοι τώρα μαθηματών θα έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν τα μαθήματα αυτά στην πλατφόρμα και επίσης θα μπορέσουν να έρθουν σε επαφή με δικηγόρους στις διάφορες χώρες. Επίσης θα έχουν τη δυνατότητα να ανεβάσουν εκπαιδευτικό υλικό. Και τώρα όσον αφορά τη διαβίου μάθηση το 2000. 16, ε, το CCB δημοσίευσε μία περίληψη για τη διαβίωμαθήση ε, στα ε, κράτη-μέλη του CCB. Έχουμε 19 πλήρη μέλη τα οποία υποστηρίζουν τη διαβίωμαθήση και στις περισσότερες εξ αυτών των χαρών το καθεστώς αυτό εισήχθη τα τελευταία 15 χρόνια. 12 πλήρη μέλη δεν έχουν υποχρεωτικό καθεστώς διαβίου κατάρτισης, όμως σε όλες αυτές τις χώρες υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, όπως για παράδειγμα ε, στην Αυστρία, στο καταστατικό εισαγγελέων προβλέπεται στο κεφάλαιο 10,6 η υποχρέωση του δικηγόρου να συνεχίζει να εκπαιδεύεται, να μορφώνεται. Και ε, έτσι λοιπόν ένας ε, μη καταρτισμένος ε, δικηγόρος με τους νόμους που αλλάζουν δεν θα είναι καλά ενημερωμένος και θα, κάνει, θα δημιουργήσει προβλήματα στον πελάτη του. Ένα μέλος, η Γεωργία, έχει υποχρεωτικό καθεστώς κατάρτισης και τουλάχιστον ένα, η Χοντούδουρα δεν έχει κανένα. είχα την ευκαιρία να με ε, ε, προσκαλέσουν δύο φορές στην Τυφλίδα και είδα με τα ίδια μου τα μάτια το πόσο ε, η περιοχή εκεί, Αζερβαϊτσάν, Γεωργία, υποστηρίζουν την διαβίου κατάρτιση των δικηγόρων χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Και για αυτόν τον λόγο υποστηρίζω πάντοτε σε όλους ε, τους ε, ειδικού ε, της Επιτροπής Εκπαίδευσης να συμμετέχουν στις συναντήσεις μας. Δεν είναι εύκολο για τις χώρες του Κάφκασου λόγω, λόγω των οικονομικών δυσκολιών να ε, παρευρίσκονται στις συναντήσεις μας, όμως συνήθως ε, στις Ολομέλειες, ε, η επόμενη θα είναι το Μάιο στο Εδιμβούργο, όλα τα μέλη θα συμμετάσχουν στην Επιτροπή. Στις περισσότερες χώρες τώρα το εύρος μετράται σε ώρες, διδακτικές μονάδες, παρόλο που σε ορισμένες χώρες μετράται ακόμα και σε μέρες. Ο, το μέσο όρος, ο μέσος όρος εκτείνεται στις 40 ε, ώρες ε, οι διδακτικές μονάδες και οι περισσότερες χώρες έχουν επιλέξει ε, τακτικό έλεγχο το οποίο σημαίνει ότι οι δικηγόροι υποχρεούνται να καταθέσουν μια αναφορά στον δικηγορικό σόλογο για την, για την εκπαίδευση που έλεγαν σε αιτήσια βάση σε ορισμένα κράτη-μέλη γίνονται τυχαίοι έλεγχοι, το οποίο σημαίνει ότι μονάχα ένας αριθμός ε, ε, δικηγορικών γραφείων και δικηγορών εξετάζονται. Υπάρχουν κράτη-μέλη επίσης τα οποία κάνουν ε, τακτικούς και τυχαίους έλεγχους. Ποιες είναι τώρα οι κυρώσεις για την έλλειψη συνεχιζούν διαβίου κατάρτισης. Υπάρχουν πειθαρχικές και μη πειθαρχικές. Οι πειθαρχικές αφορούν την προειδοποίηση μέχρι και την αποβολή από το δικηγορικό σύλλογο, ε, ενώ το μη πειθαρχικό είναι η πληρωμή κάποιου προστίμου. Εν κατακλείδη λοιπόν, Μία από τι μεγαλύτερε προσπάθειε τη Εκπαιδευτική Επιτροπή είναι να συνεργαστεί με την Επιτροπή, με την Κομισιόν για την συλλογή ε, ε, δεδομένων σε ετήσιο επίπεδο σχετικά με το κατά πόσο το Ευρωπαϊκό Δίκαιο συμμετέχει σε, αυτές τις, σε αυτά τα μαθήματα και σε αυτέ τι αναφορέ. Θα πρέπει να ομολογήσουμε όμως ότι έχουμε μια έλλειψη δεδομένων από τους ιδιωτικούς παρόχους εκπαίδευσης. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο πρόβλημα οργανώνοντας ε, ε, κατά τα τέλη της χρονιάς ε, το Δεκέμβριο στις Βρυξέλλες ένα συνέδριο για την για την εκπαίδευση δικηγόρων, τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες όπου θα συναντηθούν τόσο ή ε, ε, τα ε, θεσμικά όσο και τα ιδιωτικά προγράμματα κατάρτισης για να δείξουμε πόσο σημαντικό είναι να συλλέξουμε όλα αυτά τα δεδομένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. ευχαριστώ. Και τελευταία ομιλήτρια είναι η κυρία Ριμπέρο Τέλ, ε, η οποία προέρχεται από το Λουξεμβούργο, από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και θα μας ε, μιλήσει για την κατάρτιση του δικαστικού προσωπικού και των δικαστικών επιμελητών ε, σε ευρωπαϊκό επίπεδο και γιατί αυτή η κατάρτιση είναι σημαντική για να εργάζονται κατάλληλα οι άνθρωποι αυτοί. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ευκαιρία που μου δίνετε να μιλήσω σήμερα για το τι κάναμε στο Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης και να σας μιλήσω για την κατάρτιση του δικαστικού προσωπικού και των δικαστικών επιμελητών. Καταρχήν θα ήθελα να πω δύο λόγια για το πρώτο σχέδιο, για το πρώτο project. Θεωρούμε ότι αυτή η μελέτη είναι πολύ σημαντική γιατί ήταν η πρώτη φορά που είχαμε την ευκαιρία να δούμε ακριβώς και να έχουμε αριθμητικά στοιχεία για το πόσοι είναι οι άνθρωποι αυτοί, οι δικαστικοί επιμελητές και το δικαστικό προσωπικό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ουσιαστικά ε, χαρτογραφήσαμε τις κατηγορίες του δικαστικού προσωπικού και μπορέσαμε να έχουμε πάνω από 100 fact sheets με πάρα πολλές πληροφορίες ε, που δεν μπορούσαμε να προσθέσουμε φυσικά στην έκθεση αυτή. Και δεν μπορούσαμε να το κάνουμε επειδή επικύλαν ε, οι κατηγορίες ε, για να κάνουμε συγκρίσεις μεταξύ των κρατών μελών. Επειδή ο λόγος και το παιδί εφαρμογής του πρώτου project ήταν να καταρτήσουμε να θεσπίσουμε την κατάρτιση στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Έτσι λοιπόν είχαμε θέσει την ερώτηση αν το δικαστικό προσωπικό υποχρεούνταν να έχει νομικές σπουδές ή όχι και πώς ε, κινεί το στην πορεία. Έτσι λοιπόν, τι κάναμε εδώ. Προτείναμε τρεις κατηγορίες και θεωρήσαμε ότι είναι λειτουργήμα που σχετίζεται με τη διαχείριση και τη δίκηση των δικαστηρίων. Έχουμε την γενική διοίκηση, ε, παραδείγματο χάρη, ανθρώπου που εργάζονται στην ηλεκτρονική δικαιοσύνη, στην, ε, στην πληροφορική. Ιτηρούν βιβλία. Δεύτερη κατηγορία, το αποκαλούμε ε, δικαστικό λειτουργήμα Παραδείγματο χάρη όπως ε, η παράδοση εγγράφων, η παροχή βοήθειας ε, σε δικαστές ε, και δικαστικές ή δικονομικές αποφάσεις σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και έχουμε και τις δικονομικές λειτουργίες, δηλαδή διασυνοριακή συνεργασία σε, αστικέ αστικές, εμπορικές, ποινικέ υποθέσεις κτλ. Έτσι λοιπόν με αυτά τα δεδομένα η μελέτη μας έδειξε ότι οι πτυχές του ευρωπαϊκού δικαίου κρύβονται μέσα σε ένα εθνικό θέμα. Όλοι οι συμμετέχοντες ε, ε, ανέφεραν την ανάγκη της συνορικής συνεργασίας και για ενισχυμένες αρμοδιότητες στις ε, ευρωπαϊκές διαδικασίες που προκύπτουν κυρίως στον ποινικό τομέα από τα ευρωπαϊκά νομοθετήματα. Έτσι λοιπόν στις συστάσεις που μπορούσαμε να παράξουμε αυτό το πρώτο σχέδιο είναι εξή. Πρέπει να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση των πτυχών του ευρωπαϊκού δικαίου. Πρέπει να πούμε ότι το δικαστικό προσωπικό συνήθως, ε, αν και ε, προσλαμβάνονται για να δουλέψουν σε ένα δικαστήριο, ακόμη και αν δεν έχουν νομικές σπουδές, μερικές φορές ε, πρέπει να μπορούν να εξηγούν στους πολίτες γιατί έρχονται στο δικαστήριο και πρέπει να δίνουν αυτές τις πληροφορίες. Αυτό είναι το καθήκον τους μερικές φορές. Γι' αυτό θέλουν περισσότερες πληροφορίες ακόμη και αν καθημερινά δεν έρχονται σε επαφή με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Προς το τέλος αυτής της ε, πρώτης μεγάλης μελέτης είχαμε και κάποιες ε, προτάσεις πάρα πολύ σημαντικές το να διασφαλίσουμε την κατάρτιση για όλο το δικαστικό προσωπικό. Όλοι συμφωνήσαμε ότι το να αναπτύξουμε εργαλεία ηλεκτρονικής μάθησης θα ήταν μια εξαιρετική λύση. Το να αξιολογούμε τους εκπαιδευτές και να αναπτύσσουμε ε, ουσιαστικά ε, κάποια μαθήματα που θα είναι επικεντρωμένα στην πρακτική. Δηλαδή θα μπορούσαμε να έχουμε προσωμιώσεις ρόλων ε, στους οποίους πρέπει να μπαίνουν γιατί πολλές φορές πρέπει να συνομιλήσουν με τους πολίτες και ενίοτε δεν έχουν πάρα πολλές πληροφορίες για το πώς να συμπληρώσουν ε, παραδείγματος χάρη ε, τα έντυπα. Έτσι λοιπόν να έχουμε καλύτερη διασυνοριακή συνεργασία και αυτό στρατηγικό στόχο για όλους τους παρόχους κατάρτισης. Και κατόπιν με αυτές τις προτάσεις έχουμε την ευκαιρία και εμείς συνεργαστήκαμε με την ε, ΆΙΠΑ, με το Υπουργείο Δικαιοσύνης ε, στην Πορτογαλία και με άλλους φορείς ε, σε άλλες χώρες. Στείλαμε την αίτηση για μια επιχορήγηση για να μπορέσουμε ουσιαστικά να αναλάβουμε αυτό το project κατάρτισης για τους δικαστικούς επιμελητές. Τι προτείνουμε μία γλωσσική κατάρτιση, μία επαγγελματική προσφορά και ήταν πολύ ενδιαφέρον να καταλάβουμε το εξής. Ήταν αυτή η πρώτη φορά που οι άνθρωποι αυτοί συναντήθηκαν μεταξύ τους και εκεί μπόρεσαν να καταλάβουν πώς εργάζονται ε, με τα ίδια μέσα. Ενίοτε δεν έχουν ούτε καν κατευθυντήριες γραμμές για τα πώς να συμπληρώσουν ε, τα έντυπα. Έτσι λοιπόν, Είχαμε αυτή την εμπειρία, ανταλλαγή πρόσωπο με πρόσωπο και είμαι σίγουρη ότι αυτή η επιχορήγηση, τώρα οδεύουμε προς το τέλος, θα προσιάσουμε την τελική έκθεση, ε, ουσιαστικά τι κάναμε, κάναμε εκπαίδευση των εκπαιδευτών, Το πρώτο είχε να κάνει με δικαστικέ συνεργασίε σε αστικέ και εμπορικέ υποθέσει και το δεύτερο σε οικογενειακέ υποθέσει και ποινικέ υποθέσει. Είχαμε 41 συμμετέχοντε. Και τα αποτελέσματα ήταν πάρα πολύ καλά. 19 από τους συμμετέχοντες που απάντησαν στα ερωτηματολόγια πιστεύουν ότι πλήρως ε, πέτυχαν τους στόχους και το 15% μπόρεσε να πετύχει το στόχο του ως 75%. Και άλλο ένα αριθμητικό στοιχείο για αυτό το project. Όταν ρωτήθηκαν αν η γνώση που κέρδισαν κατά το σεμινάριο οδήγησε σε υιοθέτηση νέων προσεγγίσεων, οι περισσότεροι είπαν ναι, 69%. Η απάντηση στην ερώτηση για το αν η γνώση που κερδίθηκε οδήγησε στη βελτίωση των επιδόσεων, το 70% απάντησε ναι, 72% συγγνώμη, και τέλος, οι συμμετέχοντες ε, ουσιαστικά ενημέρωσαν και τους εκπαιδευτές για το τι μαθαίνουν, τι θέλουν να μάθουν και επίσης η ιδέα είναι να διαδίδεται η γνώση. Γι' αυτό σε αυτό το consortium μπορέσαμε να δημιουργήσουμε μια ηλεκτρονική πλατφόρμα όπου έχουμε μαθήματα στα αγγλικά, αλλά υπάρχει και δυνατότητα πρόσβασης σε μία κατάρτιση για το πώς μπορούν να εφαρμόζονται οι κανονισμοί στον τομέα του αστικού δικαίου, του εμπορικού δικαίου, αλλά και κατευθυντήρες γραμμές για τη συμπλήρωση των εντύπων και τα παραρτήματα, των παραρτημάτων. Και συμπερασματικά σε ό,τι αφορά αυτή την επιχορήγηση. Οι συστάσεις και προτάσεις για βελτιώσεις του σεμιναρίου, αλλά και για τη συνεργασία είναι το εξή. Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτή τη φόρμουλα, να έχουμε και αυτή την κατάρτιση πρόσωπο με πρόσωπο, αλλά να έχουμε και μεικτή μάθηση. Ουσιαστικά το προσωπικό θα μπορούσε να έχει πρόσβαση σε ηλεκτρονική μάθηση, αλλά στη συνέχεια όταν πρέπει να έχουμε προσωμιώσει, θα πρέπει να έχουμε κατάρτιση πρόσωπο με πρόσωπο. Θέλουν να ενισχύσουν τη συνεργασία και ίσως υπάρχει και ένα εμπόδιο γλωσσικής φύσεως. Γι' αυτό το λόγο ξεκινάμε με την πρώτη επιχορήγηση δράσης που να δώσει τη δυνατότητα σε ορισμένους από αυτούς να έλθουν και να έχουν καλύτερη πρόσβαση σε αγγλική ορολογία. Βέβαια αυτό δεν ε, σημαίνει ότι ε, θα πρέπει να συνδεθούν όπως έγινε στην Τιζόν ε, ή αλλού και υπήρχαν και ομάδες που μιλούσαν πορτογαλικά ή γαλλικά. ίσως θα πρέπει να βρουν και μια κοινή γλώσσα, ένα τρόπο επικοινωνίας. Λεχθέντος αυτούς. Η ΆΙΠΑ με την ίδια ομάδα μου υποβάλλει μια νέα πρόταση το Νοέμβριο, πέρσι δηλαδή το κάναμε, ίσως θα έχουμε καλά νέα σύντομα και θα θέλαμε να ενισχύσουμε αυτή τη συνεργασία και να έχουμε τη δυνατότητα το δικαστικό προσωπικό και οι δικαστικοί επιμελητές να λαμβάνουν κατάρτιση, γιατί φυσικά και αυτό είναι τμήμα ε, του έργου μας. Μπορούμε να δούμε τώρα ολόκληρη την εικόνα. Και φυσικά το δικαστικό προσωπικό και οι δικαστικοί επιμελητές είναι πολύ σημαντικοί για πρόσβαση σε μια καλύτερη δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστούμε πολύ. Ο χρόνος πιέζει. Έχουμε τώρα τρεις πολύ σύντομες παρεμβάσεις. Και βέβαια καλό θα ήταν να μπορέσουμε να έχουμε και κάποιες ερωτήσεις. Ένα λεπτό καθένας για τις σύντομες παρεμβάσεις παρακαλώ. Γιατί 4 και 30 πρέπει να ολοκληρώσουμε. Πρόκειται για τον δόκτωρα Χέζελ πρώτα απ' όλα. Ραουλ Μάτελ και Βάντερ Πύρ. Έτσι εσεί οι τρει. Είσαστε εδώ και τρει. Ωραία. Μπορείτε να τα καταφέρετε σε ένα λεπτό παρακαλώ. Άντε, δύο λεπτά. στι τέσσερι και μισή δεν έχουμε πια διερμηνία. Βλέπετε κάποιοι μίλησαν 15 λεπτά. Εγώ θα προσπαθήσω σε ένα λεπτό να κάνω την ερώτησή μου. Εντάξει, τότε. Όχι, ας ακούσουμε. Α, και εσείς κυρία Μακαβέ έχετε μια ερώτηση. Ωραία, στο τέλος. Πρώτα απ' όλα, ο Δόκτωρ Χάζελ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δύο λεπτά είναι δύσκολο, όπως καταλαβαίνετε. Οπότε, μην χάσω χρόνο. Ευχαριστώ για την πρόσκληση, βέβαια και θέλω να σας ε, βοηθήσω στις συζητήσεις που κάνετε στην Επιτροπή σας, εξηγώντας σας τι κάνουμε εμείς την πράξη, ποιες είναι οι αρχές, ε, σε ποιε έννοιε βασιζόμαστε. Έχουμε τρει κατηγορίε. Προγράμματα για βέλτιστε πρακτικέ, συνεχόμενα προγράμματα και νέε πρωτοβουλίε. Από τις βέλτιστες αυτές πρακτικές κατά το παρελθόν θα αναφέρω δύο μία που έγινε για δικηγόρους και νομικούς στο λεγόμενο Defense Council και το άλλο έχει να κάνει με δοκιμές που κάναμε σε διάφορες χώρες για την περίπτωση του Defense Council. Η προσέγγιση μας ήταν ότι υπήρχαν ομάδες από διάφορες χώρες τέτοιων αμυντικών συμβουλίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συζήτησαν πως τα νομικά μέσα που έχουμε όσον αφορά τη συνεργασία σε ποινικά ζητήματα λειτουργεί. Και μετά ε, συγκεντρώθηκαν σε εθνικές ομάδες προσπαθώντας να εφαρμόσουν τις αρχές αυτές σε συγκεκριμένη ομολογία, συγκεκριμένες ε, περιπτώσεις. Το άλλο ήταν ένα πρόγραμμα για 600 συμμετέχοντες από όλες τις χώρες μέλη. Δεν μπορώ να σας πω τις λεπτομέρειες, πάντως το αποτέλεσμα ήταν ότι οι περιπτώσεις που εξετάστηκαν στα πλαίσια αυτού του προγράμματος δόθηκαν δωρεάν, μπήκαν στην ιστοσελίδα και σε πολλές γλώσσες μάλιστα, γιατί όπως είπαμε και πριν το γλωσσικό μπορεί να είναι εμπόδιο, είναι ένα πρόβλημα. Εδώ λοιπόν βλέπετε τις διάφορες περιπτώσεις, βλέπετε το, τις δωρεάν πληροφορίες που βάλαμε εμείς για τις περιπτώσεις αυτές και όποιος θέλει μπορεί να έχει πρόσβαση και να ενημερωθεί για πολλά και διάφορα ζητήματα. Ένα άλλο στοιχείο που θέλω επίσης να σας αναφέρω είναι μια σειρά διαφόρων μέτρων κατάρτισης που πήραμε εδώ και χρόνια που επικεντρώνονται σε ζητήματα κατά των διακρίσεων. την έννοια αυτή κάθε χρόνο 600 καταρτιζόμενοι συμμετέχουν από όλα τα κράτη-μέλη και τέλος ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον project ε, με τη CCB είναι το θέμα ε, των διαφορών για τους δικηγόρους. Εδώ στοχεύουμε σε νέους νομικούς οι οποίοι έρχονται σε επαφή με συναδέλφους από άλλες χώρες. Κατόπιν έχουμε τα νέα project, δεν θα μπω σε λεπτομέρεια εδώ, απλώς ήθελα να τονίσω ότι όλα αυτά τα project που βρίσκεται στα έγγραφα έχουν χρηματοδοτηθεί ή συγχρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα δικαιοσύνης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θέλω να σας δείξω τι γίνεται εδώ με τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε. Δεν ήθελα να σας πιέσω έτσι, αλλά πάση περιπτώσει ευχαριστώ που κάνατε την παρουσίασή σας έστω και σε τόσο λίγο χρονικό διάστημα. Τώρα. Ο Ράουλ Ραντόι, επίση ένα-δύο λεπτά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία που δίνετε στου συμβολογράφου τη Ευρώπη να σα παρουσιάσουν τη δικιά του περίπτωση στα πλαίσια τη επιμόρφωση. Κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί και εμείς εφαρμόζουμε το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Όπως είπε και η κυρία Σούντερ νωρίτερα, διαπιστώνουμε ότι στην έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 2016, 35% των συμβολογράφων συμμετείχαν σε επιμορφωτικά σεμινάρια. Τα δύο προγράμματα Ευρώπη για συμβολογράφους και συμβολογράφοι για την Ευρώπη ισχύουν από το 2013 και έχουν προχωρήσει μέχρι και φέτος. 3.000 συμβολιογράφοι εποφελούνται από επιμόρφωση στο ευρωπαϊκό δίκαιο από 22 χώρε μέλη. Όλες τις χώρες μέλη, δηλαδή που έχουν ε, συστήματα αστικού δικαίου, καλύπτουν όλε μα τι χώρε. 26 σεμινάρια οργανώθηκαν σε 14 διαφορετικέ χώρε. Τρει ε, περιπτώσει είχαν ε, με πολλέ εθνικότητες οργανώθηκαν, δηλαδή από διαφορετικέ χώρε συγχρόνω. Προσφέραμε υλικό και βιβλία μετά από κάθε σειρά σεμιναρίων, 8 βίντεο που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας. Έχουμε επίσης συνεργασία με πανεπιστήμια, σημαντικά πανεπιστήμια, εδώ δίνουν καθηγητές, νομικούς, ομιλητές στα σεμινάρια. Συνεργαζόμαστε και με την ΕΙΠΑ από το Λουξεμβούργο για την αξιολόγηση των σεμιναρίων αυτών. Όλη αυτή η δουλειά δεν θα γινόταν φυσικά χωρίς την πολύτιμη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γι' αυτό θέλω δημόσια να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μας για την στήριξη και την εξαίρετη συνεργασία που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η επιτυχία μας κάνει να κοιτάμε ακόμα πιο μακριά τώρα και να προσπαθούμε να σκεφτούμε ιδέες για άλλα θέματα που έχουν ε, να κάνουν ε, με τους γάμους, το ότι ισχύει δηλαδή για τα καθεστώτα αυτά στις διάφορες χώρες. Έχουμε καιρό να προετοιμάσουμε τους βολογράφους. Πρώτα ευχαριστώ. Βάλτε πύρ. την τώρα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και εμείς από τη δικιά μας την πλευρά θέλουμε να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας που μας δίνεται τη δυνατότητα να σχολιάσουμε για τη συνεργασία που έχουμε με τα δικαστήρια. Υπάρχει υποχρέωση για την υπηρεσία μας να προσφέρει επιμόρφωση σε όλους όσοι συμμετέχουν σε δικαστήρια. Και η επιμόρφωση αυτή είναι υψηλού επίπεδου και έχει ως στόχο να δημιουργήσει μεγαλύτερη σύγκληση στις αποφάσεις που λαμβάνονται και στις πρακτικές που εφαρμόζονται και που έχουν νομικό χαρακτήρα. Ετοιμάζουμε λοιπόν σειρά μαθημάτων με συμμετοχή εκπροσώπων των δικαστηρίων, των δικαστικών από όλες τις χώρες μέλη και στο δίκτυο αυτό συμμετέχουν και οργανώσεις όπως είναι η Διεθνής Οργάνωση Δικαστών που ασχολούνται με υποθέσεις ασύλου και άλλες οργανώσεις που έχουν να κάνουν με την ομολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Συμβούλια κλπ. Περιλαμβάνονται και 8 οργανώσεις, το EG10 και η ΕΡΑ και υπάρχουν και εθνικά σώματα επιμόρφωσης που συμμετέχουν στο δίκτυό μας. Όλες οι δραστηριότητες που γίνονται στο δίκτυο αυτό γίνονται με πλήρη σεβασμό της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης και πρέπει να αναγνωρίσουμε τον ιδιαίτερο ρόλο που παίζουν δικαστές και τον εκτελεστικό χαρακτήρα της ΕΑΣΟ. Έχουμε 8 κύκλους μαθημάτων που πηγαίνουν από την εισαγωγή στη διεθνή προστασία, την επικουρική ε, συνεργασία το 15 σε τον αποκλεισμό, αποδείξεις, αξιοπιστία, διαδικασίες ασύλου και για του χρόνου προβλέπουμε κάτι για το θέμα της χώρας προέλευσης. Είναι σημαντικό λοιπόν να ξέρουμε ότι όλα αυτά κυκλοφορούν στη συνέχεια. Υπάρχουν κάποιοι επιμορφωτές οι οποίοι είναι δεκαστές οι ίδιοι και επανέρχονται και άλλοι συνάδελφοι πηγαίνουν σε διάφορες χώρες αλλά και σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης πηγαίνουν και παρουσιάζουν τα πορίσματα των μαθημάτων αυτών. Την επόμενη εβδομάδα για παράδειγμα πηγαίνουμε στην Ελλάδα σε διάφορα δικαστήρια που εξετάζουν προσφυγές και έτσι μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας όχι μόνο μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και εκτός, για παράδειγμα την Ισία και Μαρόκο. Ευχαριστώ πολύ και καθώς ε, φτάνουμε στο τέλος αυτού του εργαστηρίου θα ήθελα να ρωτήσω αν ε, τα μέλη έχουν ε, κάποια τελευταία σύντομα ε, σχόλια. Ρικίτ παρακαλώ σύντομη. Ε, ευχαριστώ. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι εκτιμώ το γεγονός ότι ε, κάναμε αυτό το εργαστήριο. Ε, θα ήθελα να κάνω κάποια σχόλια και να είμαι σύντομη. Πρώτα απ' όλα, ελπίζω ότι ε, καθότι κάθε ευρωπαϊκή νομοθεσία γίνεται αργά ή γρήγορα εθνική νομοθεσία, θέλω να ελπίζω ότι θα γίνεται ε, και κομμάτι της εκπαίδευσης. Ε, όμως νομίζω ότι είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η βάση ε, για, τον, ε, για έναν εθνικό νόμο είναι ένας ευρωπαϊκός νόμος, διότι όταν το ζήτημα αφορά ε, διασυνοριακές υποθέσεις ποινικού ή οικογενειακού δικαίου, τότε θα πρέπει να γνωρίζουμε, να εξετάσουμε τη βάση. Επίσης, πιστεύω ότι είναι σημαντικό ε, ότι όταν όσον αφορά την αύξηση της ε, κατάρτισης ατόμων θα πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι προφανώς υπάρχει έλλειψη χρόνου για τους ε, δικαστές και τους δικηγόρους ε, να κάνουν αυτή την κατάρτιση και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να ασκήσουμε πίεση σε τουλάχιστον κάποια από τα κράτη-μέλη μας να έχουν αρκετό προσωπικό ούτως ώστε να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο και υπάρχει και συζήτηση σχετικά με το πώς μπορούμε να ελέγχουμε τη μόνιμη κατάρτιση. Ε, κάτι ακόμα το οποίο δεν ξέρω αν αναφέρθηκε είναι ότι είναι σημαντικό να ε, αυξήσουμε την ενημέρωση σχετικά με, ε, με ποια είναι η ενημέρωση των πολιτών και η γνώση των πολιτών για τους πολίτες. Έχουμε για παράδειγμα ε, πληροφορίες από πολίτες να υπάρχει ενημέρωση από την πλευρά του Υπουργείου Δικαιοσύνης στα σχολεία για να υπάρχει αυτή η γνώση. Το χρησιμοποιούν αυτό για παράδειγμα στο πλαίσιο του σχολικού εκβοβισμού μέσω του ίντερνετ να πηγαίνουν δηλαδή στα σχολεία όχι μονάχα από ηθικό επίπεδο αλλά και από ένα νομικό επίπεδο ποια είναι τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις σου και τι μπορεί να σου συμβεί ως θύμα αλλά και ως θήτης όταν ε, κάνεις ε, σχολικό εκφοβισμό μέσω του ίντερνετ ή άλλους τομείς. Ένα τελευταίο σημείο το, σημείο το οποίο συζητήσαμε ε, κατά τα διαδικαστικά δικαιώματα στην Ευρώπη νομίζω ότι θα πρέπει να αυξήσουμε τα δικονομικά ε, μέτρα είναι ότι θα πρέπει να έχουμε ένα είδος ε, πρόγραμμα Εράσμους όπου ο καθένας θα, θα μπορεί ε, να έχει να συμμετάχει σε αυτό όταν μιλάμε για νομικούς και είναι σημαντικό να ενισχύσουμε τις προσπάθειές μας για να υπάρξει μια πρόοδο σε αυτό το τομέα. Σας ευχαριστούμε πολύ, Μπριγκίτ. Η κυρία Πεσερέλ. Ευχαριστώ δύο λόγια. Και εγώ έχω νομική κατάρτιση. Άκουσα τα προβλήματά σας, τα γλωσσικά και πράγματι νομίζω ότι είναι θεμελιώδες γιατί νομίζω ότι μέσω της γλώσσας, μέσω του πώς χρησιμοποιεί κανείς τη γλώσσα, σχηματίζει τη σκέψη του και εγώ λυπάμαι γιατί έχει αμερικανοποιηθεί το δικαίωμα μας ε, και πραγματικά διαλέγετε τα αγγλικά και αυτό πραγματικά ε, με κάνει να ανατριχιάζω. Τώρα, με το σύστημα πληροφορικής ε, δεν μπορούμε να προβλέψουμε να έχουμε ελάχιστα δεδομένα έτσι ώστε κάθε ώρα να ανταποκρίνεται σε κάτι. Ενοχλήθηκα πάρα πολύ όταν μελετούσαμε το δίκαιο δημιουργού και στα γαλλικά έχει μεταφραστεί copyright. Και για μένα αυτό είναι ακριβώς το αντίθετο από τα δικαιώματα του δημιουργού. Από τα δικαιώματα του δημιουργού. Λοιπόν, οι ακροάσεις είναι πάντοτε πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και σας ευχαριστώ για όλη τη δουλειά που κάνατε. Thank Σας ευχαριστούμε που θέσατε και αυτό το γλωσσικό θέμα. Είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Πολλοί μιλούν κακά αγγλικά και φυσικά δεν αρμόζει στα νομικά επαγγέλματα. Οι δικηγόροι είναι πάρα πολύ ευφύς άνθρωποι και πρέπει να αγωνίζονται σε μια γλώσσα που δεν είναι η δική τους. Και όταν ε, εγώ ήρθα εδώ υπήρχαν τα γαλλικά. Τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η κυρία Μακοβέη, παρακαλώ, που έχει εργαστεί και για το φάκελο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και τους προσκεκλημένους μας Χαίρομαι που βλέπω και τους φίλους μας από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Έχω συνεργαστεί 10 χρόνια με το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ε, κάναμε κάποιες αποστολές με το Συμβούλιο της Ευρώπης για ανθρώπινα δικαιώματα και τη μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος. Τώρα, εγώ προέρχομαι από μια πρώην χώρα. Έπρεπε να μεταρρυθμίσουμε το δικαστικό σύστημα μετά το 1990 και ήταν πολύ δύσκολη αυτή η μεταρρύθμιση και είδα ότι όλες οι άλλες χώρες που ήθελαν να μας βοηθήσουν παρουσίασαν την κατάρτιση. Κανένα δεν ενδιαφερόταν για την κατάρτιση τότε. Οι χειρότεροι ε, δικαστές εστάλησαν για κατάρτιση και οι καλύτεροι κρατήθηκαν για να δουλέψουν στο δικαστήριο γιατί την κατάρτιση θεωρούσαν κάτι άχρηστο. Άλλαξαν τα πράγματα κάπως με το πέρασμα του χρόνου. Όμως και τώρα, όσο μιλάμε, υπάρχουν κράτη-μέλη που έχουν βασικές ανάγκες. Δεν έχουν του χάρη υπολογιστέ, δεν έχουν διαδίκτυο. Και νομίζω ότι αυτό προέχει της κατάρτισης. Γιατί θα μπορούσαν ε, να πιστούν να ακολουθήσουν την κατάρτιση και μετά να πάνε σε ένα δικαστήριο που δεν έχουν αυτό τον εξοπλισμό. Στι περισσότερε μετακομμουνιστικέ χώρε ε, δεν ε, μπορείς ε, παραδείγματος χάρη καν ε, να δακτυλογραφήσεις την κατάθεση ενός μάρτυρα. Εξακολουθεί να καταγράφεται με το χέρι και έτσι λοιπόν δεν γίνεται καταγραφή λέξη προς λέξη. Έτσι λοιπόν, εγώ νομίζω ότι αν έχουμε κονδύλια, καταρχήν πριν από την κατάρτιση αυτά πρέπει να κάνουμε, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να είναι χρήσιμη η κατάρτιση. Και κάτι τελευταίο. Η διαχείριση των δικαστηρίων είναι κάτι διαφορετικό. Ένα άλλο πρόβλημα το οποίο θα πρέπει να λύσουμε σε αυτές τις νέες δημοκρατίες. Τώρα, αν ε, κάνετε κατάρτιση για την ενοποίηση της ε, νομολογίας, εγώ δεν θεωρώ ότι υπάρχει ξεκάθαρο σύνορο μεταξύ του πυρωτικού δικαίου και του συστήματος common law. Βλέπουμε το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ευρωπαϊκών Δικαιωμάτων, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο, χρησιμοποιούν ομολογία τα δικαστήρια αυτά. Αυτό είναι σωστό, γιατί δεν χρειάζεται οι άνθρωποι να πάνε στο δικαστήριο ε, σαν να αγοράζουν λαχείο. Πρέπει να είναι προβλέψιμη δικαιοσύνη. Αν ε, έχω υπογράψει μια σύμβαση, πρέπει να ξέρω ποια είναι η ανάλογη νομολογία οι δικαστές λένε είμαστε αμερόληπτοι και η ενοποίηση της νομολογίας βλάπτει, ουσιαστικά πλήττει την αμεροληψία μας. Αυτό όμως είναι λάθος. Δεν νομίζω ότι οι Βρετανοί δικαστές αισθάνονται λιγότερο ανεξάρτητοι αφού έχουν αυτό το σύστημα common law. Επίσης, πρέπει η δικαιοσύνη να είναι προβλέψιμη κατευθυντηρίες γραμμές, ε, παραδείγματο χάρη, για ποινέ, όλα αυτά τα πράγματα τα χρειαζόμαστε. Έτσι λοιπόν η ενοποίηση της νομολογίας ε, είναι πάρα πολύ σημαντική στα πλαίσια της κατάρτιση. Τα δύο διεθνή δικαστήρια που έχουμε στην Ευρώπη εργάζονται καλύτερα βάσει νομολογίας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Μακοβέη. Ευχαριστώ τα μέλη που παρευρέθησαν εδώ. Ευχαριστώ και την κυρία Ντελβό και θέλω να ευχαριστήσω και τους συναδέλφους ε, στη Γιούρη. Ξέρω ότι υπάρχουν και πάρα πολλές παρασκηνιακές ε, συνεδριάσεις. Εγώ συνειδητοποίησα ότι είχαμε πάρα πολλές ε, συνεδριάσεις. Ζητήσατε το λόγο. Σαν πολιτικός συμπεριφέρεστε συμπερασματικά. Δυστυχώς, η επερχόμενη συνεδρίαση κατάρτισης που πρέπει να γίνει το Δεκέμβριο θα γίνει μόνο στην αγγλική γλώσσα, γιατί θέλαμε να μειώσουμε το κόστος της μετάφρασης. Μάλιστα. Έχουμε εδώ Ιταλούς, Πορτογάλους και όλοι μιλάτε πάρα πολύ καλά αγγλικά. Βέβαια έχετε δίκιο σε αυτό που είπατε πρέπει να δούμε και το θέμα της ακρίβειας των νομικών όρων. Έχετε και κάτι άλλο να πείτε, αστιεύεστε. Για ένα δευτερόλεπτο μπορώ. Δεν θέλετε να γίνετε πολιτική; όχι. Θα μιλήσω γαλλικά για να ικανοποιηθεί η κυρία Μπερζερόν και θέλω να απευθυνθώ στην κυρία Μακοβέη. σα ευχαριστώ πολύ για το σχόλιο που κάνατε στο τέλος σε σχέση με την εναρμόνιση της νομολογίας σε εθνικό επίπεδο. Αυτό δεν είναι ένα θέμα ομογενοποίησης. Ε, η κατάρτιση για τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι ένα από τα εργαλεία για να εξασφαλίσουμε την υλοποίηση των ευρωπαϊκών κανόνων σε εθνικό επίπεδο. Υπάρχουν βέβαια και πολλά άλλα εργαλεία και το Συμβούλιο της Ευρώπης εργάζεται πάρα πολύ σε όλα αυτά τα θέματα εναρμόνισης της νομολογίας σε εθνικό επίπεδο για να εξασφαλίσουμε ότι οι εθνικές δικαιοδοσίες ερμηνεύουν με συνεκτικό τρόπο και την νομολογία του ΕΔΑΔ αλλά και την νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ που το είπατε αυτά. ουσιαστικά ε, δεν θα ήθελα τώρα να αναφέρουμε και σε διάφορες ευαίσθητες επιτυχίες με τις οποίες ασχολείται η Άσο. Πάντως είναι καλό να έχουμε κάποια συζήτηση όταν γίνεται το πρόγραμμα με ένα συγκεκριμένο τρόπο. Ευχαριστώ τους εμπειρογνώμονες για τις παρουσιάσεις ε, που ήταν και παθιασμένες. Παρόλο που δεν είχαμε μεγάλη συμμετοχή, εμείς θεωρούμε ότι ήταν πάρα πολύ σημαντική αυτή η συζήτηση για να κατανοήσουμε και το στόχο αλλά και την ποιότητα της κατάρτισης. Είχαμε εξαιρετικές παρουσιάσεις σήμερα και οι δύο επιτροπές μας ε, θα προωθήσουν τα διδάγματα αυτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για αυτές τις ουσιαστικές παρουσιάσεις. Σας ευχαριστώ όλους για το χρόνο σας σήμερα και εσύ είμαστε σε στενή επικοινωνία. Ε, αν η Κομισιόν παρουσιάσει και νέες προτάσεις. Να είστε σε επαφή μαζί μας σας παρακαλώ. Σας ευχαριστώ.